και θα ήθελα να ευχαριστήσω λοιπόν την εισηγήτρια και επιστρέφω τώρα τα δύο λεπτά που σας είχα κλέψει από την προηγούμενη παρέμβαση. Ευχαριστώ. Θαυμάσια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Επίτροπε. Ολοκληρώνω τη συζήτηση του θέματος αυτός της διάταξης και περνάμε στο επόμενο σημείο. Την έκθεση Νικολάη σχετικά με τη θέση των γυναικών στου πολέμου. Και θα ήθελα να δώσω την εισηγήτρια για τέσσερα λεπτά το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσω να καλύψω σε τέσσερα λεπτά όλη την έκθεση. Όμως, να σας πω μερικά θέματα που θα θεωρώ πάρα πολύ σημαντικά. Πρόκειται για κάποια έκθεση η οποία έρχεται στην σωστή χρονική στιγμή. Ε, έχουμε τις πρωτόγονες κοινωνίες οι οποίες χρησιμοποίησαν τον βιασμό ως όπλο, ως μέσο πολέμου. Επομένως πρόκειται για ένα θέμα τώρα το οποίο είναι καυτό τη καθής επικαιρότητας και έχει πάρα πολύ σοβαρές κοινωνικές ε, συνέπειες και επηρεάζει βεβαίως και την πολιτική των ε, κρατών. Α, κοιτάξτε τι έγινε στον πόλεμο του Κονγκό. Εκεί είχαμε 16 βιασμούς ανά ημέρα. Πρόκειται για μια μάστιγα η οποία με τίποτα δεν έχει αντιμετωπιστεί. Αυτή η έκθεση έχει ξεκαθαρίσει ότι το θέμα θα πρέπει να το δούμε και σαν θέμα ισότητας φίλων και ισότητας ευκαιριών. Θα πρέπει οι γυναίκες και άντρες να το αντιμετωπίσουν χέρι-χέρι και να προλαμβάνουν κάποιες ε, συγκρούσεις. Θα πρέπει επίσης μετά τις συγκρούσεις και τους πολέμου να πηγαίνουμε σε ε, ανασυγκρότηση. Θα πρέπει επομένως να ληφθούν αποτελεσματικά βήματα ούτως ώστε ε, να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο γιατί έχουμε μόνο 10 κρατη τα οποία έχουν πρόγραμμα, έχουν πολιτική. Έχουμε άλλα πέντε κρατημέλη τα οποία δουλεύουν προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά όλοι οι άλλοι υστερούν πάρα πολύ όσον αφορά τις προσπάθειες αυτές. Θα πρέπει επομένω να δούμε πώς θα μπορέσει να βοηθήσει και η υπηρεσία εξωτερική δράση, ούτω ώστε να ε, προβληθεί περισσότερο το πρόβλημα, το οποίο είναι καυτό. Έχουμε κάποιες ε, αντιπροσωπείες οι οποίες έχουν εμπλακεί και ασχολούνται με το πώς θα καλυφθούν οι γυναίκες, πώς θα, θα βελτιώσουμε και αυτό το ψήφισμα, και έτσι να μπορέσουμε να ε, έχουμε μια ειρήνη η οποία θα διαρκέσει. Να μην υπάρχει ατιμωρησία. κάτι το οποίο ισχύει σήμερα. Θα πρέπει επίσης να επιλαμβάνει των σχετικών περιπτώσεων το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Άρα θα πρέπει να αναζητήσουμε τις νομικές μεθόδους που θα οδηγήσουν στην τιμωρία των ενόχων, οι οποίοι και αυτοί με τη σειρά τους θα πρέπει να παραπεμφθούν στο δικαστήριο. Αντιθέτως δεν θα πρέπει τα θύματα να ενοχοποιούνται και να σταματήσει η ατιμορρησία που σοβεί σήμερα. Θα πρέπει επομένω ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά ε, και ο ΙΑ να κάνει περισσότερα. Έχουμε δεδομένο το ψήφισμα 1960 και επομένως με τέτοιες κοινές προσπάθειες το φαινόμενο αυτό να καταπολεμηθεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επιδείξει στεναρή στάση για να προσφέρει βοήθεια και ασφάλεια στις γυναίκες. Θα πρέπει το, πρόβλημα αυτό να δοθεί από πλευρά ισότητα των φίλων. Να υπάρχει περισσότερη αξιοκρατία. Θα πρέπει επίσης να λαμβάνουν και ηγετικέ θέσεις και στις ενοπλές δυνάμεις οι γυναίκες οπότε όπω προείπα δεν μπόρεσα να καλύψω όλα όσα θα ήθελα μέσα σε τόσο λίγο χρόνο Όμω αυτό το οποίο θέλω είναι να ευχαριστήσω του σκιώδει ηγητέ όλων των πολιτικών ομάδων. Ευχαριστώ. Ε, σας ευχαριστώ κύριε ηγητρία. Πάλι έχουμε περισσότερους που έχουν ζητήσει το λόγο στο ΚΑΣΕΑΙ από τη χρόνο έχουμε. Θα δώσουμε λοιπόν κατά προτεραιότητα το λόγο σε εκείνους που δεν έχουν μιλήσει ακόμα και να προσθέσουμε να έχουμε και μια ισορροπία φίλων. Στην Α Ματέρα, ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, χαίρομαι πάρα πολύ για την ε, εκλογή σας ως Αντιπροέδρου. Σας συγχαίρω και θα ήθελα να συγχαρώ επίσης τη Α Νικολάη για την έκθεση αυτή που είναι πάρα πολύ καλή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των γυναικών, ιδίως εκείνων των γυναικών οι οποίες ε, σε μια κατάσταση πολέμου ε, εμπλέκονται και δεσμεύονται γιατί βλέπουν ε, συχνά μαζικούς βιασμούς και άλλα τέτοια παρόμοια γεγονότα που θεωρούνται ότι είναι μια κοινή πρακτική πολέμου και είναι τα πρώτα θέματα οι γυναίκες Αυτά όλα έχουν και, και επιπτώσει στην υγεία, αλλά και στην ψυχολογία των γυναικών και των οικογένειών τους. Θα πρέπει αυτές τις καταστάσεις να τις ε, ε, καταδικάζουμε πολύ πιο αυστηρά και δεν θα πρέπει να περνάνε ατιμόρυτες οι πράξεις αυτές. Δικαιοσύνη είναι πάρα πολύ σημαντική και αυτό σημαίνει ότι θα ήταν καλό στη δικασία της ε, την ηρευτική να συμμετέχουν και γυναίκες για να μπορέσουν να ενταχθούν σε αυτές τις πρακτικές. Ευχαριστώ, συνάδελφε. Η κυρία Φιλαζίκα Βαβένοβα έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τις τελευταίες δεκαετίες ε, δεν επιτύχαμε παρά μικρή πρόοδο σε αυτό το τομέα. Πολλές φορές υιοθέθηκαν κάποιες ε, ποσοστώσεις και αυξήθηκε το ποσοστό των γυναικών στους διάφορους οργανισμούς. Παρ' όλα αυτά η συμμετοχή των γυναικών διαπραγματεύσει για ειρήνη είναι τη τάξη του 10%. Αλλά οι γυναίκε παίζουν σημαντικό ρόλο <clears throat> όσον αφορά την, ε, ε, τις πολιτικές αναλλαγές και οι τοπικές εκεί οι γυναίκες μπορούν να διαπραγματευτούν με τις τοπικές αρχές πολύ καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο. Τα δικαιώματα μας των γυναικών δεν ε, θεωρούν τόσο σημαντικά, θεωρούν δεύτερης ε, διαλογής αν θέλετε και οι τοπικές συνήθειες ε, αιτιολογούν ε, υποτίθεται την συμπεριφορά προς τις γυναίκες. Θα πρέπει λοιπόν αυτό όλο να τα λάβουμε υπόψη μας. Γιατί στη δημιουργία ειρήνης όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέει πρόεδρος. Ο κύριος Ζωμέρο Ερβέντα έχει το λόγο. Yeah, thank you. Ευχαριστώ πρόεδρε. Νομίζω ότι το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ λεπτό. Βεβαίως και είναι σημαντικός ο ρόλος των γυναικών ως θύματα των πολέμων. Αλλά επίσης είναι σοβαρό το θέμα και λόγω του ρόλου που μπορούν να, πέσουν, να παίξουν οι γυναίκες όσον αφορά την ειρήνευση, την ανασυγκρότηση των ε, κοινωνιών και έτσι να αλλάξει αυτός ο δρόμος που οδηγεί τα κράτη στους, στον πόλεμο. Άρα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το όσα ε, έχει πει ο ΙΕ στο 18-20, στο 18-25, τα ψηφίσματα εκείνα. Επίσης ε, έχουμε συγκεκριμένο εκπρόσωπο, συγκεκριμένο ε, αξιωματούχο που ασχολείται με αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένω, πρόκειται μια ευκαιρία. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το θέμα να το θεωρήσει ψήφι προτεραιότητα στην εξωτερική πολιτική στις σχετικές μας ε, δραστηριότητες. Όχι, δεν είναι έλασον το θέμα. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία που δεν πρέπει να την χάσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, συνάδελφε. Η κυρία Τσέσκοβα, τώρα για ένα λεπτό. Ε, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Πρόκειται για φρικτά αποτρόπια εγκλήματα κατά γυναικών, κατά κοριτσιών που γίνονται στου πολέμου. Επομένω, θα πρέπει κάτι να γίνει, πρέπει να καθούν περισσότερε προσπάθειε. πότε για την σεξουαλική βία, ομαδική βιασμή, δουλεμπόριο, διάφοροι τρόποι ε, ε σεξουαλικών εγκλημάτων που γίνονται με ευκαιρία ε, του πολέμου που γίνονται πάντω στον κόσμο. Αυτό είναι απαράδεκτο, είναι προσβολή τη ανώμη αξιοπρέπεια και επομένω, ε, όπω πολύ σωστά τα λένε οι συγκητές θα πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι είναι μια εγκληματική δραστηριότητα. Αυτή η δραστηριότητα θα πρέπει να προσαχθεί με τις δικαιοσύνες με μηδενική ανοχή. Γιατί όσα γίνονται στους πολέμους, για όσα γίνονται στα προσφύγων, άρα θα πρέπει να δούμε πώς θα αναβαθμιστεί ο ρόλος των γυναικών σε επίπεδο πολιτικού διαλόγου, σε, όσον αφορά τις ε, σχετικές ε, ε, στρατιωτικές και μη στρατιωτικές αποστολές. Ευχαριστώ, συνάδελφε. Δύο μιλητές μπορούμε ακόμα να πάρουμε για το ΚΑΤΔΙ. Η κυρία Νεντέλη Τσέβατα. Ένα λεπτό παρακαλώ. Merci, Monsieur le Pendant les deux premières guerres mondiales, les... Ευχαριστώ, Στους δύο πρώτους ε, παγκόσμιους πολέμους οι γυναίκες έχαναν τους γιους και τους άντρες τους ε, στο μέτωπο. Σήμερα όμως είναι άμεσα θύματα. Βιάζονται, σκοτώνονται, είναι ιδιαίτερα ευάλωτες. Ε, χαίρομαι που επιτέλους το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκφράζεται ώστε η βία κατά των γυναικών στον πόλεμο να θεωρηθεί σαν έγκλημα πολέμου. Γι' αυτό είμαστε ευγνώμονες προς την εισηγήτρια την κυρία Νικολάη. Υπάρχουν ε, βέβαια οι επιπτώσεις στην υγεία αλλά και στην ψυχολογία των γυναικών αυτών. Επίσης υπάρχουν ε, σημαντικές επιπτώσεις πάνω στους άντρες που δεν μπόρεσαν να αντιταχθούν, δεν μπόρεσαν να προστατεύσουν τις γυναίκες τους και τις κόρες τους. Και στα παιδιά που βλέπουν τι διαμείβεται, τι γίνεται, τι συμβαίνει. Οι γυναίκες θα πρέπει να παίξουν ρόλο στην επίλυση των ε, διαμαχών στην αναζήτηση της ε, ειρήνης. Και τέλος θεωρώ ότι η Ένωσή μας στα κέρδη δεν είχε ειδικό εκπρόσωπο για την, υγεία, την, την γυναίκα, συγγνώμη, την ασφάλεια και την ειρήνη. Δεν ξέρω. Μπορούμε να δημιουργήσουμε μια τέτοια θέση και αν είναι, πότε. Ευχαριστώ. Τελευταίο ομιλητή, ο κύριος Λουάν. Ένα λεπτό. Και η Υποπιτροπή Ασφαλείας και Αμήνης ασχολήθηκε με αυτά τα εγκλήματα κατά των γυναικών και είχαμε προσπάθειες για καταπολέμηση της ατιμορρησίας που είναι απαράδεκτη. Δυστυχώς η βία των γυναικών χρησιμοποιείται ως τακτική, πολεμική και δυστυχώς σε πολλές περιπτώσεις έχουμε βιασμούς, εγκλήματα τέτοια τα οποία δεν καταγγελώνται καν. Θα πρέπει η υπηρεσία εξωτερικής υπηρεσίας να ορίσει έναν ειδικό παρατηρητή, επόπτη για το τι γίνεται στις πολεμικές ζώνες και έτσι να υπάρξει κάποια προσπάθεια βελτίωσης της κατάστασης. Σας ευχαριστώ. Σας είδα κυρία Συνεβέρη το θέμα, δεν έχουμε όμως ε, απεριόριστο χρόνο, αλλά έχουμε και περιορισμένο αριθμό ομιλητών. Δεν λυπούμε πάρα πολύ. Εάν μπορούσαμε θα δίναμε το λόγο σε όλους. Δυστυχώ δεν είναι δυνατόν. Από την άλλη μεριά θα πρέπει όμως να προχωρήσουμε. Ίσως κύριε Στρίφνερ, εντάξει, θα σας δώσω το λόγο, αλλά λάβετε υπόψη ότι ε, στο μέλλον δεν θα μπορεί να ακολουθούμε την, την τακτική ότι όλοι μιλάνε όσοι θέλουν. Αλλά μια που το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό, θα ήθελα να σα δώσω το λόγο για ένα λεπτό πριν δώσουμε το λόγο στην κυρία Επίτροπο. Σα ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, και θα Το, το θέμα τη σεξουαλική βία που χρησιμοποιείται σαν όπλο πολέμου είναι ένα πρόβλημα σε όλο τον κόσμο. Εμεί πολλέ φορέ έχουμε ασχοληθεί με το θέμα αυτό που επιδεινώνεται ιδίω στην Ανατολή τη ε, δημοκρατίας του Κονγκό. Εγώ πήγα στο, Νότιο Κιβούλ πριν από λίγο χρόνο. Είδα πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση και πόσο σημαντικέ είναι οι φυσικέ και ψυχολογικέ επιπτώσει στι γυναίκε και στα κορίτσια έναντι αυτή τη βία, η αναπροβολική και η σεξουαλική υγεία θα πρέπει να είναι ένα θέμα που θα μα απασχολήσει. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει κεντρικό και σημασία στα θέματα αυτά και στην προστασία των γυναικών στον τομέα τη σεξουαλικότητα στον πόλεμο. Είναι ένα έγκλημα, ένα έγκλημα πολέμου αυτό. Γιατί η γυναίκα δεν είναι μέσω πολέμου, δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, συνάδελφε. Πέντε λεπτά εξ ονόματο τη Επιτροπή, η κυρία Γεωργίευα έχει το λόγο. Thank you, Mr. President. Ευχαριστώ. Αξιότιμοι βουλευτές, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω με πάσα ειλικρίνεια την κυρία Νικολάη, την συγγήτριά μας. Ευχαριστώ επίσης που ακολουθεί αυτό το θέμα ένα παρεμφερέ ζήτημα που μα απασχολεί εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη βία δηλαδή κατά των γυναικών. Ο ρόλος των γυναικών έχει ιδιαίτερη σημασία για μας, ε, κυρίως ο ρόλος τους ε, στις, δραστηριότητες, στις ειρηνευτικές δραστηριότητες μέσα από το ψήφισμα 1325 του ΟΗΕ και άλλων ε, συναφών ψηφίσματων. Θέλουμε να έχουμε μία ολοκληρωμένη προσέγγιση σε όλα τα όργανα εξωτερικής δράσης, σε, όλα τα, σε όλες τις πολιτικές και όλα τα προγράμματα. Το 2008 ενέκρινε η Επιτροπή μια σφαιρική προσέγγιση για τα ψηφίσματα 13-25 και 18 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΙΕ, ώστε να καλύψουμε όλα τα θέματα, όλα στις φάσεις ε, πριν και μέσα, μετά την ε, διένεξη. Ε, στο 13-25 μιλάμε για τη συμμετοχή, την προστασία των γυναικών και την πρόληψη της βίας εναντίον των γυναικών. Θα ήθελα εδώ να μιλήσω για τη χρηματοδότηση εν συντομία Έχουμε το όργανο για τη σταθερότητα, το Ευρωπαϊκό Μέσο μάλλον για τη σταθερότητα. Πρόκειται για ένα εργαλείο κλειδί που μας επιτρέπει να σταθεροποιήσουμε τα μέτρα οικοδόμησης ικανοτήτων και ειρηνευτικών δραστηριοτήτων, προστατεύοντας και τα δικαιώματα των γυναικών καθώς και των πλέον ευπαθών ομάδων, δηλαδή τα παιδιά, οι γυναίκες, οι ανάπηροι, οι ηλικιωμένοι στα πλαίσια της δράσης μου ε, ως Επίτροπος ε, ε, για την Ανθρωπιστική Δράση ε, προσπαθούμε σε κάθε πολιτική μας να βοηθούμε τις ε, γυναίκες μέσα από αυτό το ευρωπαϊκό μέσο. Επίσης, έχουμε προγράμματα που ονομάζονται Cash for Work με τριτά ε, εναντίον εργασίας, για τη εργασία μάλλον, για να βοηθήσουμε τις γυναίκες, όπως παραδείγματο χάρη στο Κονγκό. Εγώ έμεινα εκεί τρεις εβδομάδες και πραγματικά ο βασικός στόχος μου θα είναι και το αντικείμενο της έκθεσής σας, δηλαδή προστασία των γυναικών να σταματήσει ο βιασμός των γυναικών που χρησιμοποιείται ως εργαλείο πολέμου. Ε, το φαινόμενο παρατηρείται σε πάνω από 70 χώρες ε, και 200 εκατομμύρια ευρώ επενδύθηκαν ε, στα τέλη του 2009 εξ αρχές του 2010 στις περισσότερες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας περάσω στην κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Οι περισσότερες επιχειρησιακές αποστολές ε, και για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για την πρόθεση ε, της ισότητας των δικαιωμάτων των δύο φύλων έχουμε τρεις διαφορετικές υποενότητες στα πλαίσια πάντοτε της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας ε, θα οριστικοποιηθούν στα τέλη του 2012. Συνεργαζόμαστε στενά επίσης με το στρατιωτικό προσωπικό για να υπάρχει μια κοινή ε, προσέγγιση για όλες τις ανθρωπιστικές ε, διαστάσεις των διενέξεων και με ποιο τρόπο οι διενέξεις αυτές επηρεάζουν τις πιο ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες. Επίσης είναι σημαντικό εσωτερικά να δράσουμε διορίζοντας ε, γυναίκες διαμεσολαβητές ή διαπραγματευτές, διορίζοντας περισσότερες γυναίκες σε βασικά ε, καθήκοντα στην υπηρεσία εξωτερικής ε, δράσης, στα κράτη-μέλη είναι ιδιαίτερα δραστήρια στα πλαίσια του ΟΗΕ. Έχουμε εθνικά προγράμματα δράση σε 13 κράτη-μέλη. Άλλοι πάλι, όπως η Γερμανία, έχουν καταλήξει σε ειδικέ πρωτοβουλίες. Ε, για το ρόλο των γυναικών ε, στα πλαίσια της ε, ασφάλειας και της ειρήνης. Ως προς την εφαρμογή του ψηφίσματος 1325 ολοκληρώθηκε το Μάιο του 2011 μία έκθεση αξιολόγηση και φαίνεται από εκεί ότι έχουν αναλυθεί συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία των πιο ευπαθών ομάδων μεταξύ των οποίων και οι γυναίκες. Μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τις προσπάθειες που ήδη έχουμε κάνει. Όμως θα παραμείνουμε σε εγρήγορση για τις δράσεις μας σε όλα τα φόρα, σε όλες τις χώρες για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση των ενόπλων διενέξεων, για να συμμετέχουν ενεργά σε ειρηνευτικές και στη δημόσια εκπροσώπηση γυναίκες και θα ήθελα να πατήσω και στην ερώτηση σχετικά με το ότι αν εξετάζουμε το ενδεχόμενο έχουμε έναν ειδικό εκπρόσωπο. Η κάθε άστον είπατε εκπρόσωπο στο Νοέμβριο ε, ανέφερε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο διορισμού ενός ειδικού επιτρόπου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ε, προσδιορίζει, οριοθετεί τη θέση προς το παρόν. Και κλείνω ευχαριστώντας σα πραγματικά για τη σημερινή συζήτηση. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Γεωργίευα. Ολοκληρώνεται εδώ η εξέταση του θέματο. Η ψηφοφορία θα γίνει σήμερα στι 12 το μεσημέρι. Επόμενο σημείο τη σήμερα διάδεξη. Η έκθεση κυρία Ευλήν Ρέγκνερ όσον αφορά την διασυνολική μεταφορά τη έδρα εταιριών. Τέσσερα λεπτά έχει το λόγο η συγκέντρια. Παρακαλώ.